So, good morning everybody. Καλημέρα σας. Αν δεν απατώμε αρχίζουμε. Με τη γνωμοδότηση πιανού Εστεβάλ δεν είναι εδώ. Μας ζήτησε όμως να αρχίσουμε με τη δική του έκθεση. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Εμίλιο Ντελβάλε. να κάνουμε. Ποιος είναι υπεύθυνο για τον κύριο Ντελβάλε. Υπεύθυνο. Να αρχίσουμε με άλλη, αλλά μαζί ζήτησε. μαζί ζήτησε. Καλά, θα αρχίσουμε με την κυρία Σάντσες Σμιτ τότε. Θέλεις να πεις τίποτε Μαρία Θηρεσία. Ναι ή όχι. Ορίστε, ορίστε. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Σα ζητώ βέβαια να υπερψηφίσετε την έκθεσή μου με τίτλο Όθηση στου τομεί του πολιτισμού και τη δημιουργία για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση. Πολύ σημαντικό θέμα προφανώ και που συνδέεται με την πολιτιστική ταυτότητα που σήμερα συζητιέται και ενδιαφέρονται πολύ. Χαίρομαι γιατί ψηφίζουμε αυτή την έκθεση, διότι μιλάει και για το οικονομικό δυναμικό του τομέα αυτού και τις δυνατότητες του να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Πάνω από 4% του εσωτερικού του χωρίου αγαθάς του προϊόντος βασίζεται στον τομέα αυτόν. Η πολιτιστική εξαίρεση πρέπει να διατηρηθεί. Εξάλλου θα γνωρίζετε ότι τα προϊόντα μας και η κληρονομιά μας έχουν μεγάλη σημασία στο, στη διεθνή σκηνή και πρέπει να τα προωθήσουμε και να τα προστατεύσουμε. Τρεις είναι οι κύριοι άξονες να τους βοηθήσουμε τον τομέα να περάσει στο ψηφιακό και να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και τρίτον να γίνει μια μελέτη για τις ε, θετικές επιπτώσεις στην οικονομία του τομέα αυτού. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία και την στήριξή σας. Α, σας ευχαριστούμε. Αρχίζουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Η 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 41 Ψήφος κατά συνείδηση, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε τώρα στην 45. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46. Υπέρ, η 47. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 ε, υπέρ κατά αποχές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 Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην άλλη σελίδα η 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το υπόλοιπο το υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ για την 79. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε παρακαλώ για την 97 έκλεισε η ψηφοφορία απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική, μισό λεπτό, συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100, μάλλον η συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 130 υπέρ κατά κατά αποχές ε, εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε 31 Vote is 21 zu 8 angenommen εγκρίνεται 132 133 και 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μισό λεπτό 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 145 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 147 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος 147. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. εγκρίνεται. 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 151 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 151. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Μισό λεπτό. Πάλι για την 159 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 162 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε παρακαλώ για την 164. Έκλεισε η ψηφοφορία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 αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 173 ε, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μισό λεπτό 175 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85-84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 14 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. 14 λοιπόν ψηφίζουμε για την 14. Έκλεισε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 15 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Vote closed. 16 zu 13 angenommen. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Μισό λεπτό λάθος έκανα. Α, συγγνώμη λέει η πρόεδρος. Στο 21, για το 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 25. Μα το προηγούμενο απορρίφθηκε μισό λεπτό. 23 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ ψηφίζουμε έκλεισε η ψηφοφορία 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την 29. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται.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 η 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 37 ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πληρώνουμε, ε, ψηφίζουμε τώρα για το σύνολο από το 1 μέχρι το 8 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Και ε, τελική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ. The vote is closed. zu 0 bei 4 Enthaltungen. Συγχαρητήρια λοιπόν στη Μαρή Τερέζ. Ευχαριστούμε. So, now we come to Mendes del Valle. Menendez del Valle. Τώρα Μενέντες del Έχετε τίποτε να μας πείτε. Όχι. Μάλιστα σας κατευχαριστούμε. Μίλησα χθε πολύ, δεν χρειάζεται και τώρα. Α, χθε ήταν ένα άλλο θέμα. Τέλο πάντων. Λοιπόν, μπείτε ζερ. Λοιπόν, η 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 34 υπέρ κατά Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την 34. Έκλεισε η ψηφοφορία. 13. Απορρίπτεται. Η 34. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. 19 προς 10. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται, 37 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 39 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την 39. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 40 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 ε, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ κατά αποχές μισό λεπτό ξανά 57 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 ήταν 60. 62 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 62. Έκλεισε η ψηφορία. 64 υπέρ κατά αποχές υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 2 εγκρίνεται, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 ή 80 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 82 ε, υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Η 3 και 85 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 89, υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 και 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 5 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την 5. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 21 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 28 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την 28. Έκλεισε η ψηφοφορία. 29 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία Ψηφίσουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ψηφίστηκε, υπερψηφίστηκε η ε, εισήγηση, η έκθεση. κύριος Αλφονσί. Ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Απλώ να πω ότι η έκθεση αυτή αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα και αφορά την πολιτιστική πολυμορφία. Πιστεύουμε ότι σήμερα και σε διεθνέ επίπεδο είναι κάτι πολύ σημαντικό και η θέση της Ευρώπης αξίζει μόνο αν είναι παραδειγματική. Ενίοτε είναι, αλλά όχι πάντοτε και έχει καθορίσει πρότυπα όπως ο Ευρωπαϊκός Χάρτης ε, των κλωστών ε, και εγώ ε, σήμερα πρέπει να δηλώσω ότι λυπάμαι που η χώρα μου, η Γαλλία δεν έχει επικυρώσει αυτή τη χάρτα, με συγχωρείτε. Αντωνία κάνε κάτι για μένα σε παρακαλώ. Βλέπετε, πάντοτε την κατάλληλη στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, θα είτε για αυτό το θέμα, ενίοτε πολιτικά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι εδώ ομόφωνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να συμφωνήσουμε για το ότι πρέπει να κάνουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για τις γλώσσες και για την ευρωπαϊκή κληρονομιά που είναι υπό εξαφάνιση και όλοι πρέπει να διαφυλάξουμε αυτή την κληρονομιά. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους γιατί υπάρχουν πολλέ ε, τροπολογίε που δείχνουν ότι ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για αυτό το θέμα και εσείς Πρόεδρε και συντονιστέ. Ε, ε, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που επιτρέψατε τη σύνταξη αυτή τη έκθεση και φυσικά όλες οι ανταλλαγέ απόψεων ήταν ιδιαίτερα καρποφόρε. Ευχαριστώ. Αρχίζουμε λοιπόν. Συμβιβαστική 4. Περκατά. Υπέρ, κατά, 75, ψηφίζουμε για την 75. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Αν ε, λιγάκι βοηθήσετε κι εσείς μπορούμε να ξεκονομήσουμε χρόνο. 76 και 77 μαζί, υπέρ κατά αποχές ε, ε, ελέγχουμε παρακαλώ για την 78 ε, έκλεισε η ψηφοφορία εγκρίνεται 77 υπέρ όχι πάμε στην 80 80 υπέρ κατά αποχές ε, ψηφίζουμε παρακαλώ για την 80 έκλεισε η ψηφοφορία Απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ψηφίζουμε παρακαλώ για την 85. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται, η 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112, 112 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές ψηφίζουμε. Έκλεισε ψηφοφορία. 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 126 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 31 και τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε παρακαλώ. Εγκρίθηκε 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 138 υπέρ κατά ε, αποχές εγκρίνεται, 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται, 146 υπέρ κατά ε, αποχές, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την ε, προφορική τοπολογία 8 και την 146 έκλεισε η ψηφοφορία. «149». 166 και 167 απορρίφθηκε, προφορική 9 και 148 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 150 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Έκλεισε η ψηφοφορία. 151 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 153 υπέρ μάλλον 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153... 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 163 και 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές Είμαστε στην 168 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Έκλεισε η ψηφοφορία. 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λάθος έκανα λέει η πρόεδρος. Λάθος έκανα προφανώς. Συμβαστική 1. Δίκιο έχετε. Και τώρα πάμε στην 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 19 και 20 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Η 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 24, 25, 24 αποσύρθηκε, για την 26 ψηφίσαμε, εγκρίθηκε, για την 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 33 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε παρακαλώ για την 33. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 39 και η 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την 47. Έκλεισε ψηφοφορία εγκρίνεται η 4 και 48 υπέρ κατά αποχές απορρίτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 7 και η 55 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την 55. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 58 υπέρ κατά... Α, ξέχασα την 57. Με συγχωρείτε. Ψηφίζουμε για την 57 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 57. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, η 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 5 η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 7 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος, ψηφίζουμε παρακαλώ για την 7. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε για την 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Για την 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ, για την 12, 12 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ψηφίζουμε παρακαλώ The vote is closed 30 zu 0 oh Alfonsi congratulations Συγχαρητήρια και σας ευχαριστούμε που το ζητήσατε αυτό. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σας. Στην ε, αρχή, όταν ξεκίνησε η αυτή η ιστορία, ποτέ δεν πίστευα ότι θα έχουμε αυτή την έκβαση. Το ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτό. Ερχόμαστε στην έκθεση Παπα-Νικολά, εφαρμογή της Στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νεολαία. Γιώργο, θες να πεις κάτι? Just thank all colleagues. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τους και οδησηγητές και φυσικά τη γραμματεία. Let us Να ξεκινήσουμε λοιπόν. γιατί 47 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται, 48 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 58 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται, η 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 61 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται, 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 85 υπέρ κατά Κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 94 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 97 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 105, 106, 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 120 υπέρ κατά αποχές υπέρ λοιπόν κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 121. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος. 121. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 122. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 123. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 126 υπέρ κατά αποχές απορριτέται, 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίζουμε παρακαλώ για την 137 Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 και 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 144 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 148 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 153 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 154 υπέρ κατά αποχές εγκρι... απορρίπτεται, 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μισό λεπτό, ξανά. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ κατά αποχές αποχές απορρίπτεται, 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 172 υπέρ κατά αποχές, μισό λεπτό, κάτι πάει καλά, μισό λεπτό, επαναλαμβάνω λέει πρόεδρος, 171 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, νομίζω έκανα λάθος λέει πρόεδρος, έκλεισε η ψηφοφορία. ήθελα να ξέρω ότι συμφωνείς ε, μαζί μου, γιατί είσαι ο καλύτερος ε, ε, στα θέματα ψηφοφορίας, αλλά μόνο σε αυτά, τέλος πάντων. Λοιπόν, ε, 173 υπέρ. Κα... Η δύο δεν έχει αποσυρθεί. Non, non, non. Non, 73 η 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 3 Λάθος είχα κάνει. 4 παρακαλώ. Η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 7 Μα την ψηφίσαμε. Η οκτώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 9 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 9. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 12 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 18 υπέρ κατά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 κατά αποχές απορρίπτεται, η 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στις ε, τροπολογίες Επιτροπής Απασχόλησης. Για τις πρώτες τέσσερις, να ψηφίσουμε για τις τέσσερις για την ABC και 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, και την 2 υπέρ κατά αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την 2 έκλεισε η ψηφοφορία απορρίπτεται η 3 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται η 4, η 5, 4 και η 5 από κοινού υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται η 6 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ για την 6. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 8 να ψηφίσουμε από την 8 μέχρι την 13. Όχι. 8 υπέρ κατά αποχές και πάλι λοιπόν ψηφίζουμε για την 8, για την 8 έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και πάλι λοιπόν ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 10. Έκλεισε η ψηφοφορία, απορρίπτεται. Για την 11. Υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 11. Ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και η 11 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Μα ψηφίσαμε για αυτή. Δεν το 11 and now 12. I, Συγγνώμη λέει πρόεδρο, συγγνώμη για την 12 ψηφίζουμε. Έκλεισε η ψηφοφορία. απορρίπτεται. Η 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οι τροπολογίε τη επιτροπή Περιφερειών τώρα. Η 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, η 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 7 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται, η 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 9 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται, η 10 υπέρ κατά αποχές γκρίνεται, η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, για όσους ε, με ακούγαν, ε, Ρεγγί, ε, εσείς που κάθεστε πίσω, είναι η Περιφερειακή Επιτροπή η οποία κατέθεσε τροπολογίες επί των οποίων ψηφίσαμε και προηγουμένως ε, ψηφίσαμε για την ΕΜΠΛ που είναι η ε, Επιτροπή Απασχόλησης. Ξέρετε τα λέμε εδώ με ακρονίμια για να προχωράμε πιο γρήγορα, να κερδίζουμε χρόνο. Ψηφίζουμε λοιπόν, έκλεισε η ψηφοφορία. Μπράβο, Γιώργο. Συγχαρητήρια. So, what do we have now? Helga. So, we come to the last and the final. Φτάνουμε στην τελευταία ψηφοφορία. Έχουμε πάρα πολλές τροπολογίες, περισσότερες ίσως και από όλες τις υπόλοιπες εκθέσεις μαζί. Λοιπόν, η κυρία Τρίπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Ντόρις, πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους και για την αποφασιστικότητά τους να βελτιώσουν την οδηγία. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ε, που προσπαθήσαμε να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Πολύ γενικά νομίζω ότι έχουμε την πλειοψηφία για να μιλήσουμε ε, για ε, την συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων και όχι για εταιρείε. Ε, δεν είμαστε κατά του ανταγωνισμού, αλλά θέλουμε να έχουμε δίκαιους κανόνες για τον ανταγωνισμό. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως να έχουμε και το ίδιο πνεύμα σε ό,τι αφορά ε, τη συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό θα το βρούμε και σε αυτή την οδηγία. Εδώ έχουμε την ίδια ιδέα σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή ε, ότι οι CMOs και οι άλλοι ανεξάρτητοι φορείς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό έδαφος θα πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Ε, μιλάμε για την ακριβή διανομή για το θέμα της προσβασιμότητας της πληροφορίας, αλλά δεν θέλουμε να θέσουμε σε κίνδυνο τα ιδιωτικά δεδομένα. Έτσι λοιπόν και πάλι εδώ μιλάμε για την κατάλληλη ισορροπία. Πολύ γενικά μιλούμε για τα, ε, το να έχουν περισσότερα δικαιώματα τα μέλη και αυτό σημαίνει ελεύθερες άδειε για, μη, ε, την μη εμπορικού σκοπού, αλλά επίσης ε, διαφυλάσσουμε και τσιμός για την πολιτιστική πολυμορφία και φυσικά κάτι τέτοιο το χρειαζόμαστε ιδιαίτερα στο ψηφιακό περιβάλλον. Και Επομένως, μιλάμε για περισσότερα δικαιώματα για καλύτερη διαχείριση των CMOs και ξέρω ότι ήταν σκληρή η δουλειά μερικές φορές, αλλά ελπίζω τώρα να βρούμε μια καλή λύση έτσι ώστε και η Επιτροπή στη συνέχεια ε, του πολιτισμού να μπορεί να διαδραματίσει έναν ισχυρό ρόλο ενάντια των άλλων επιτροπών. Μάλιστα, ευχαριστώ Χέλγα, να ξεκινήσουμε. 81. και 82 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τώρα πάμε στην 15, στην επόμενη σελίδα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο συμβασμό 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμό 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμό 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 187. Υπέρ, κατά αποχές για να το ελέγξουμε για την 187 14-15 απορρίπτεται 189 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 189 άρχεται ψηφοφορία πέρας Πέρας. 19 προς 10 εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 190. 15 προς 12 εγκρίνεται. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ κατά αποχές έλεγχους. 195. 16 προς 11 εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές για την 24 16 προς 13 εγκρίνεται. 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 203. 19 προς 10 εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές. Συγγνώμη, καταπίπτει. 26, 204 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 205 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά αποχές έλεγχος πέρας 15 προς 12 εγκρίνεται 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 215 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 216 εγκρίνεται 217 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρας. 16 προς 12 εγκρίνεται. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28 Υπέρ, κατά. Εποχές, απορρίπτεται. Συμβασμός 7, υπέρ. Κατά. Εποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. εποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το δούμε. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. 16 προς 11 εγκρίνεται. 30 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 30 πέρας Λοιπόν, πάμε, απορρίπτεται. 2,25 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 2,26 υπέρ κατά, αποχές. Για το 26 Ψηφίζουμε πέρα της ψηφοφορίες. 16 προς 13 εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Εποχές έλεγχος. Γιατί 28 πέρας. 15 προς 12 εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για την 32. Πέρας. 10 προς 19 απορρίπτεται. 2.30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος γιατί είναι 230. Πέρας. 16 προς 12 εγκρίνεται. 2.31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.42 υπέρ 2.42. Συγγνώμη, πήγα πολύ γρήγορα. Ποιο είναι υπέρ για τη 2.42. Κατά, εποχές. Να ελέγξουμε. Τη 2.43 λέει τώρα η μιλήτρια. Πέρας. 15 προς 14, απορρίπτεται. 2.44, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.45 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Γιατί είναι 2.45. Εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.46 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2.47 υπέρ, κατά, αποχές. Γιατί δύο 2.47 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 16 προς 12 εγκρίνεται. Λοιπόν, οι υπόλοιπες αποσύρονται μέχρι την 37. Υπέρ, κατά, από εγκρίνεται 37. 2.51 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 254 απορρίπτεται 255 και 256 απορρίπτεται 2.57 εγκρίνεται. 2.58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβασμός 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα, 2.74. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 2.75. Υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε. Πέρας. Ένα λεπτό. Ξέχασα να ψηφίσω. Να το ελέγξουμε παρακαλώ. Γιατί δεν το 5. Και πάλι άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Πολύ περίεργο. Κάποιος δεν ψήφισε, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Λοιπόν, 40 υπέρ κατά. 276 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 277 υπέρ κατά εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 280 απορρίπτεται. 281 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 282 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 283 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 284 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 285 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 287 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 233 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. για τη 233. Ένα λεπτό. Θέλω να ρωτήσω πόσοι από το ΕΛΚ ψήφισαν. Όχι πάρα πολύ. Κοιτάξτε, το κάνει αυτόματα το μηχάνημα. Δυστυχώς είμαστε κάπως περισσότεροι. Και, και πάλι για τη 233, αλλά το μηχάνημα μου λέει ότι έχουμε παραπάνω από όσους θα έπρεπε. No. Μου λέει είναι παραπάνω. Τώρα έχουμε 13. Κάποιος όλος ψήφισε με το ΕΛΚ, μπορεί. να σας πω κάτι. Είναι πολύ έξυπνο το μηχάνημα. Μας ε, λένε ψήφισαν παραπάνω από 12 από το ΕΛΚ ε, ή αν πάνω από 8 ή 9 από τους σοσιαλιστές. Και από τους ελεύθερους. Είναι έξυπνο το μηχάνημα λοιπόν. Πού είχαμε μείνει. Λοιπόν, είχα ανοίξει πληροφορία για τη 233. Πέρας ψηφοφορίας. 18 προς 11 απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 286 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 288 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές συγκρίνεται. 290 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 291 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 293 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 294 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2,96 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία για το 2,96 πέρας 16 προς 13 εγκρίνεται 2,97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 305 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 307 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 321 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 319 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 308 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 309 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 311 δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 212 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 313 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 315 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 316 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σας παρακαλώ σταματήστε ή να αποχωρήσετε. 16 Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξω για 416. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. 13-13. Απορρίπτεται. 13 13 απορριπτεται 317 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 318 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 320 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 322 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ξεκίνησε η ψηφοφορία, Γιώργο. Α, μάλιστα. Πέρας. 13 προς 12. 13 κατά 12 υπέρ, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά αποχές. Εγκρίνεται 325 υπέρ, κατά εποχές να ελέγξουμε για τροπολογία 325. Πέρας. Απορρίπτεται. 326 υπέρ, κατά, Εποχές απορρίπτεται. 327 υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε την 327 έρχεται ψηφορία πέρας 13-13 απορρίπτεται 328 υπέρ κατά αποχές έρχεται ψηφοφορία να ελέγξουμε πέρας 14 προς 13 εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 56 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε, άρχεται ψηφορία, πέρας, 13-13 απορρίπτεται, 3-30 υπέρ κατά Αποχές, να ελέγξουμε αρχή συμφορία. Πέρας. 22 προς 5 εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 331 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά θα συγκρίνεται, 334 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε άρχεται ψηφορία για την 334 πέρας 12-15 απορρίπτεται, τροπολογία 60 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται, 336 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 335 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 337 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε. Άρχεται ψηφορία. Πέρας. 14 12 εγκρίνεται. 338 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 339 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 340 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 341 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 342 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά όχι καταπίπτει αυτή 346 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και έχουμε ταυτόσιμες τροπολογίες. Πάμε λοιπόν στην Λοιπόν, έχουμε μέσα όπω σα είπα. Πάμε στην 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 349 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 351, έλεγχος. Για την 349 λέει μιλήτρια έλεγχος, έρχεται ψηφορία πέρας. Απορρίπτεται. 351 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Άρχεται ψηφορια Πέρας. Αντίκρουση 14 απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 352 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 353 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 354 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε στην 71 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. 356 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. 357 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται. 358 υπέρ κατά αποχέ, έλεγχο έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 16 προς 11 εγκρίνεται. 3,59 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 360 υπέρ κατά αποχές έλεγχος έρχεται ψηφορία. Για την 360 πέρας απορρίπτεται 9 προς 17. 361 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 362 υπέρ κατά αποχές, έλεγχος, άρχεται ψηφορία. Πέρας. 6 11 εγκρίνεται. 363 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Πέρας. το Λοιπόν, 364 εγκρίνεται, 365 εγκρίνεται, 366 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 367 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρας. 12-12 απορρίπτεται. 368 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος. 8 Πέρας. Απορρίπτεται. 369 υπέρ κατά. Για 369. Υπάρχει μια ερώτηση για την 368. Τι κάνουμε να ελέγξουμε. Εγκρίνεται. Ε, οπότε έχουμε φτάσει στην 369. Σωστά. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφορία για την 369. Πέρασμα. Εγκρίνεται 15-12. 370 υπέρ. Κατά. Αποχέ απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 372 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 371 υπέρ κατά αποχέ. έλεγχος αρχή ψηφορία. Πέρας. εγκρίνεται 13-14, 373 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 374 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 375 και 376 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 380 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 381 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 32 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 383 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 384 υπέρ, κατά, εγκρίνεται, 385 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 386 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 389 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 75 υπέρ κατά, όχι, μάλιστα, συγγνώμη, καταπίπτει, 88 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 76 υπέρ κατά Αποχέ απορρίπτεται 77 υπέρ κατά Αποχέ απορρίπτεται 390 υπέρ Κατά. Αποχέ. Έλεγχο. πέρας 13-12 εγκρίνεται 80 Πέρ. Συγγνώμη. Κάτι προσπέρασα. Συμβασμό 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 Συγγνώμη, 85 υπέρ. Κατά. Χες. Έλεγχος για το 85. Άρχεται η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγγνώμη. Για το 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τερπολογία 4. να ελέγξουμε. Άρχεται ψηφορία για την τροπολογία 4, πέρας. 9 προς 16 απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, Αποχέ συγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, Αποχέ συγκρίνεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχο για την 91. Πέρας. Εγκρίνεται. Να πάμε στην 95. Υπέρ, κατά, αποχέσει εγκρίνεται. 96. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 6. Υπέρ, κατά, αποχές έλεγχος. Άρχεται τη για την 6. πέρα 5 προ 12 απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά. Αποχές έλεγχος. 97 άρχεται η πέρα περας Πέρας. 14-13 απορρίπτεται. 98 υπέρ κατά. αποχέ, έλεγχο για την 98. Πέρας. 13-14 απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά εποχές έλεγχος. Αρκετά ψηφορή για την 99 πέρας. Mm. Εγκρίνεται. 100. υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 102, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός 13, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 110, υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 111, υπέρ, κατά, εποχές, απορρίπτεται. 112, υπέρ, κατά, Αποχές έλεγχος για την 112. Πέρας. 8 εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για την 113 άρχιδη ψηφορία. Πέρας. 22 προς 5, απορρίπτεται 114, υπέρ, κατά, απορρίπτεται, συμβασμός 14, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 119, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, έρχεται ψηφορία, για την 119. 13 zu 13 abgelehnt. 120 dafür, dagegen, Enthaltung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 Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Έλεξε. Εγκρίνεται 24 ψήφοι υπέρ 0 κατά 3 αποχές. Ο κύριος Καβαντά ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει άμεση σχέση με την ψηφοφορία. Θα ήθελα όμως τα πρακτικά της συνεδρίασής μας να αναφέρεται ρητά ότι μερικοί βουλευτές δεν εγκρίνουν αυτά που δήλωσε στο ΖΙΤΑ 8 ο πρόεδρος της Κομισιόν που μου φαίνονται σκανδαλώδη για δύο λόγους. Πρώτον, δεν είναι δουλειά του να κρίνει την ε, πολιτιστική εξαίρεση γιατί είναι κάτι που έχει εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Και δεύτερον, το επίθετο αντιδραστικός που χρησιμοποίησε για όσους τάσσονται υπέρ είναι σκανδαλώδες. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, τα γεγονότα απέδειξαν τον ίδιο και γι' αυτό μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Και σε αυτό συνέβαλε και το Κοινοβουλίο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το καταγράψουμε στα πρακτικά. κύριος Να πω δύο λόγια στα φιλανδικά. Η πρόθεσή μου δεν ήταν να διαταράξω τη διαδικασία της ψηφοφορίας, όμως ε, πιστεύω ότι δεν μιλάμε για fair play για στους κανόνες ε, έχουμε εδώ μια αντιπροσωπεία και όταν ε, κατά τη διάρκεια κάποιες ψηφορίες διαπίστωσα ότι είχαμε 13-14 που έρχονταν από το ΕΛΚ εγώ νόμιζα ότι ο ακριβής αριθμός ήταν 11 και νομίζω ότι έπρεπε να παρεμβούμε. Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο έξυπνο το μηχάνημα, δεν ξέρω όμως πώς διαβάζει παραδείγματος χάρη το μηχάνημα της ψήφου των φιλελευθέρων, το χάρη, όμως αυτό που με εκπλήσει είναι ότι κάποιοι όπως ο κ. Παπα-Νικολάου και άλλοι σταμάτησαν να ψηφίσουν. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι πρέπει εδώ να σεβόμαστε τους κανόνες του παιχνιδιού. Ξέρουμε πώς είμαστε εδώ από κάθε πολιτική ομάδα. Κοιτάξτε, δεν θέλω τώρα να λέω άσχημα πράγματα, αλλά δεν αισθάνομαι και τόσο άνετα. Αν δεν εκπροσωπούνται ε, όλοι εδώ, υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Γιατί ναι, ε, είναι το μηχάνημα FES, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ισότητα για όλους. Δεν πρέπει να υπάρχει κατάχρηση εξουσίας εδώ. Αυτά ήθελα να πω. Κοιτάξτε, η συσκευή δεν μπορεί να είναι δίκαιη. Η συσκευή το μόνο μπορεί να κάνει να ελέγχει και αυτή η συσκευή απλά ελέγχει πόσοι ψήφισαν του ΕΛΚ, πόσοι φιλελεύθεροι, σοσιαλιστές, οτιδήποτε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Βρήσε με όσο αλλά η συσκευή ούτε δίκαιη είναι, ούτε άδικη, κάνει μόνο τη δουλειά της. Και αυτό πάντα έτσι ήταν. Τώρα, αν δεν σε βόλευε σήμερα, πρόβλημά σου. <clears throat> Δεν ψήφισε ούτε ένας από το ΕΛΚ ε, από όσου δικαιούνταν ήταν περισσότεροι στην αίθουσα, αλλά δεν ψήφισαν. Η συσκευή δουλεύει δίκαια, σωστά. Εγώ δεν είχα ποτέ προβλήματα με τις συσκευέ. Μπορούμε να ε, πούμε στους ελεγκτέ να ελέγξουν τι μηχανές αν δουλεύουν σωστά. Δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει αυτό. τέλο πάντων. Αυτό που είπε, είναι ridiculous, ε, λέει κατά λέξη η πρόεδρο. Τι να κάνω εγώ τώρα. Εγώ προσπαθώ να είμαι πάντα δίκαιη, αλλά στις ε, ψηφορίες ούτε δίκαιη ούτε άδικη μπορώ να είμαι. Ε, Βεβαίω ελέγχω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Φοβάμαι, χάνω ότι σήμερα κοιμήθηκε στραβά. Ε, λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, στον προϋπολογισμό. Yeah. Okay. Ladies and gentlemen, Κυρίε και κύριοι, τώρα θα πρέπει να σας διαβάσω κάτι στα αγγλικά, γιατί δεν είναι εδώ ο Μόρτεν και πρέπει να σας ζητήσω να ακολουθήσετε τους κανόνες στους οποίους έχουμε συμφωνήσει. Να σας διαβάσω το κείμενο και να με ακούσετε. Δεν το κάνει τώρα το μηχάνημα, εγώ η ίδια. Λοιπόν, η Επιτροπή θα θετήσει μόνο το σχέδιο προπολογισμού για το 2014 στις 26 Ιουνίου αυτό είναι πολύ αργότερο από το συνήθως και δυστυχώς σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα για την κατάθεση τροπολογιών και για την γνωμοδότηση. Καταρχήν, ο εισηγητής μας, ο Λόκεγκαρτ, θα παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του όπου θα θέσει τις πολιτικές προτεραιότητες για τον Ιούλιο. Όμως, επειδή το προσχέδιο του προπολογισμού θα υιοθετηθεί τόσο αργά, θα διατίθεται μόνο στα αγγλικά. Πρώτον. Δεύτερον, ο κύριος Λόκερκαρτ επίσης θα παρουσιάσει τις τροπολογίες του στο προσχέδιο προϋπολογισμού και πάλι μόνο στα αγγλικά τον Ιούλιο. Και σε αυτή τη συνεδρίαση θα πρότεινα να του δώσουμε μια συγκεκριμένη εντολή όπως κάναμε πέρσι για να αποκαταστήσει τα νούμερα της Επιτροπής εκεί όπου θα δούμε περικοπές από το Συμβούλιο. Τρίτον, ε, η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι για τις 17 Ιουλίου, για τις τροπολογίες των μελών στο προσχέδιο προπολογισμού και για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις, καθώς και για το σχέδιο της γνωμοδότησης. Τέταρτον, το σχέδιο της γνωμοδότησης, τροπολογίες του εισηγητή και δικής σας τροπολογίες, όλα αυτά θα μεταφραστούν. Πέμπτο, θα ψηφίσουμε επί όλων των πτυχών της διαδικασίας προϋπολογισμού σε μία έκτακτη συνεδρίαση που θα διαρκέσει μία ώρα στις 5 Σεπτεμβρίου το πρωί. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να σταλεί σε όλους, εντάξει. Θα ψηφίσουμε λοιπόν στις 5 Σεπτεμβρίου επί όλων των πτυχών τη διαδικασία του προπολογισμού σε μια εκτακτή συνεδρίαση. Συμφωνείτε με τη διαδικασία αυτή, ελπίζω. Θα σα ε, δώσω και τα στοιχεία. Κύριε Μπελέτ, παρακαλώ. Απλώς να ελέγξω αν ε, θα υπάρξει μια συναλλαγή για τις ε, απόψεων για το θέμα αυτό. Υπάρχει μια ημερομηνία που να έχει καθοριστεί ήδη. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα αν είναι μόνο στα αγγλικά οι τροπολογίες, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα αρχής εδώ. Μόλις πέρασε, δεχτήκαμε μια έκθεση για την ε, γλωσσική ποικιλότητα και πρέπει να μπορούν οι βουλευτές να δουλεύουν στη γλώσσα τους. Θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσω ότι είναι ίσως ατυχές αυτό που έγινε και πρέπει να έχουμε τα μέσα να τα μεταφράζουμε όλα, <clears throat> ιδίως για τόσο σοβαρά θέματα όπως τον προϋπολογισμό. Μα σας είπα όλες οι τροπολογίες και οι δικές σας και του εισηγητή θα μεταφραστούν πριν ψηφίσουμε. Εν τω μεταξύ όμως υπάρχει μια δυσκολία όχι λόγω ημών. Τι να πω σας πω εγώ. Δεν μπορώ να αλλάξω τα πράγματα. Ευχαριστώ πάντως που ως αγγλόφωνοι τάσεσθε υπέρ της γλωσσικής ποικιλία. Το Συμβούλιο δεν έκανε τη δουλειά του εν καιρός. Το τέλος όμως θα μεταφραστούν όλα, μην ανησυχείτε. Τίποτε άλλο. Όχι, ερχόμαστε στο 13. Α, εχθές είχαμε το ελληνικό θέμα, το κλείσιμο της ΕΡΤ δηλαδή. Κάποιος ζήτησε να λάβει το λόγο από αυτού του θέματος σήμερα, αλλά δεν είναι εδώ. Απάντως μας αφορά όλους. Δεν ξέρω αν έχετε δει και εγώ επέκρινα πάρα πολύ αυτή την πράξη. Την κυβέρνηση δηλαδή γιατί έδρασε με τόσο ομό και βίο τρόπο. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα στις χώρες μας να κλείσει κανείς από τη μια στιγμή στην άλλη ένα σταθμό. Είναι θέμα συμπεριφοράς. Δεν μιλάω για το κατά πόσον ο σταθμός αυτός είχε υπερβολικά πολλούς εργαζόμενους, αλλά ποιος τους διόρισε, ποιος έτσι γίνεται πάντα στην Ελλάδα. Όλες οι διοικήσεις έχουν υπερβολικά πολλούς δημόσιους υπαλλήλους αλλά που δεν τους χρειάζονται. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτά χρονίζουν τα προβλήματα και η ΕΡΤ έπρεπε να μειώσει το κόστος της αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό με το κλείσιμο πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο. Αυτό ήθελα να πω. Το κάμα είδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η κυρία Ντόρις Πακ. Ε, νομίζω ότι είναι παντελώς απαράδεκτο. Ε, από τη μια στιγμή στην άλλη να τραβάει κανείς την πρίζα και να κλείνει ένα σταθμό. Χαίρομαι πάρα πολύ για την απόφαση που έλαβε εχθές το βράδυ το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε ότι η απόφαση της κυβέρνησης ε, είναι παράτυπη και ότι θα πρέπει να αρχίσει και πάλι να εκπέμπει η ΕΡΤ και ενώ θα λειτουργεί ε, μπορούν να γίνουν διάφορες σκέψεις ε, για την αναδιάθρωσή τους και το βρίσκω όλο αυτό πραγματικά πολύ κουταπώνυρο με την έννοια ότι όλοι αυτοί που προσλήφθηκαν οι ίδιοι διαμαρτύρονται παρότι πριν από κάποιους μήνες ε, είχαν πει το αντίθετο. Δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει ε, για κάποιο κόμμα, αυτό ισχύει για όλους ε, στην Ελλάδα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο το να εκφράζονται επιχειρήματα ότι αυτό το απέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω κανείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν ζήτησε να κλείσουν ραδιοτηλεπτική σταθμή. Απλά ζητήθηκαν εξοικονομήσεις κονδυλίων. είναι όμως ε, δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να κλείσει το ραδιόφωνο ή τηλεόραση γιατί καταλαβαίνετε ένα τέτοιο γεγονός ε, απλά εξάπτει τα πνεύματα στην Ελλάδα κάτι που δεν είναι επιθυμητό αυτή τη στιγμή. Ελπίζω λοιπόν στην Ελλάδα να αρχίσουν διαπραγματεύσεις να προσπαθήσουν να αναδιαρθρώσουν το ραδιόφωνο και την τηλεόραση γιατί σίγουρα δεν είναι τώρα αυτός σταθμός στην Ελλάδα όπως ε, τον ξέρουμε στη Γερμανία στην Αγγλία εγώ λοιπόν ελπίζω ότι τώρα πλέον ε, θα έχουμε έναν ε, ανεξάρτητο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό στην Ελλάδα και με συμμετοχή των ε, δημοσιογράφων ελπίζω ότι θα αναζητηθεί αυτή η διέξοδος και πιστεύω όπου οι Ευρωπαίοι μπορούν να υποστηρίξουν πρέπει να το ψάξουν. Αλλά αυτή η διαδικασία πραγματικά ήταν απαράδεκτη και προφανώς μπορεί κανείς μόνο να την ε, καταδικάσει ε, με, έμφαση. Συμφωνώ όμως, είπε η Πέτρα, και θέλω να προσθέσω δύο δεινά. Καταρχήν, Βεβαίω, το κλείσιμο της, δημόσιας, ε, της ελληνικής δημόσιας υπηρεσίας ε, μου φαίνεται πραγματικά επίθεση κατά της δημοκρατίας αλλά και μία μη αιτιολογημένη επιλογή γιατί μπορούν να υπάρξουν προβλήματα και δυσκολίες. Ναι μεν, αλλά μπορεί να γίνει ένας σχεδιασμός για μίσου του προσωπικού όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Αλλά πραγματικά η επιλογή αυτή μου φάνηκε παράδεκτη. Δεύτερον, υπήρξε ε, και ένα αίτημα από τα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά δίκτυα που ζήτησαν την ελληνική κυβέρνηση να ξανασκεφτεί το θέμα. Είναι αλήθεια ότι η Επιτροπή δεν ε, έχει καμία ευθύνη στο ότι ε, έκανε μια τέτοια ένδειξη. Αυτό θα μας έλειπε να ζητήσει κάτι τέτοιο η Τρόικα. Όμως στη δήλωση της Κομισιόν στο Στρασβούργο λέγοντας ότι είναι μια επιλογή της κυβέρνησης και δεν υπάρχει καμία υπευθυνότητα της Κομισιόν και μάλιστα επαναλαμβάνεται ο λόγος της δημόσιας υπηρεσίας ότι η Κομισιόν ε, ίσως ε, θα έπρεπε να λάβει μία δράση υποστήριξης, να επαληθεύσει αν ε, πληρούνται οι προϋποθέσεις και με κάποιο έκτακτο μέσο παρέμβασης να βρεθεί μια διαφορετική λύση. Τώρα, πέρα από την τηλεόραση, καταργείται και η φιλαρμονική και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική μοναδική την πηγή, γιατί ξέρετε ότι κλείνει η συμφωνική ορχήστρα. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή επίθεση εδώ κατά του πολιτισμού και το δικαίωμα στην πληροφορία, του δικαιώματο στην πληροφορία και νομίζω ότι πρέπει το Κοινοβούλιο να απευθύνει ένα αίτημα στην Κομισιόν για να μπορεί να βρεθεί μια συμπεφωνημένη λύση για να υπερασπιστούμε τι αρχέ που για μα δεν είναι δυνατόν να τι απομπέψουμε. Και κάτι ακόμη να προσθέσω.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 έχει πάλι μετάφραση. Ναι, τώρα δουλεύει. It's working now, German. Okay. Marco. Λοιπόν, ο Μάρκο. Κοιτάξτε, έλεγα προηγουμένως ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση όπου έχουμε απόλυτο παραλογισμό. Καταρχήν, έχουμε ένα δημόσιο ε, ραδιοτηλεοπτικό σταθμό που είναι μια ανοιχτή κλίνη. Βεβαίως ε, δεν σέβεται κανείς τη δημοκρατική διαδικασία της ενημέρωσης και της ε, συμμετοχής έτσι ώστε να γνωρίζει κανείς ε, τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει χωρίς κρατική τηλεόραση καμία δυνατότητα να έχει κανείς αντικειμενική ενημέρωση και επίσης ε, ε, δεν είναι δυνατόν και να υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες στην κοινωνία. Απ' την άλλη όμως έχουμε το εξής παράλογο. Έχουμε μία ε, τηλεόραση υδροκεφαλισμένη με προσωπικό παντελώς άχρηστο και το προσωπικό αυτό πληρωνόταν για να μην κάνει τίποτα, ουσιαστικά τίποτα. Αυτά λοιπόν είναι τα δύο θέματα τα οποία πρέπει κανείς να εξετάσει και εμεί ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς ως ευρωπαϊκός θεσμός, κυρίως ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουμε εκλεγεί άμεσα από τους πολίτες. Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι ως Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή πρέπει να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης ε, για να πούμε ε, στην Ελλάδα ενδεχομένως το πώς ε, μπορεί σε συντομότατο χρονικό διάστημα να ανασυστήσει μια κρατική τηλεόραση. Γιατί αυτό σας λέω άπλεται και της δημοκρατίας στη χώρα αυτή σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Κατόπιν τούτου πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις με πολύ μεγάλη προσοχή. Απ' την άλλη πρέπει βέβαια, όπως σας είπα, να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να δώσουμε κάποιο μέλλον σε όλους αυτούς τους πλέον άνεργους. Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι ιδιαίτερη. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνεργοι και άλλοι που δεν έχουν ε, καμία σχέση με την ΕΡΤ. Στον ιδιωτικό τομέα λυπάμαι που δεν έχουμε εδώ κάποιον Έλληνα έτσι ώστε να μας πούνε και εκείνοι ποια ε, είναι η δική τους άποψη, αλλά σας λέω ε, πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια στο βαθμό που μας αφορά όλη η υπόθεση έτσι ώστε η κρατική ραδιοτηλεόραση να ανασυσταθεί το συντομότερο ε, δυνατόν γιατί σε μια, με μια οικονομική και κοινωνική κρίση αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε πολιτική και να εκφυλιστεί σε καταστάσεις που δεν θα αρέσουν σε κανένα. Ωραία. Είναι λοιπόν ρητό το δικαστήριο, το δικαστήριο πρέπει να ξανανοίξει η ΕΡΤ. Και αυτό το θέμα πρέπει να μιλήσουμε που είναι η συμπεριφορά της κυβέρνησης που κάνει απαράδεκτα για τη δημοκρατία πράγματα. Η Χέλγα. Ευχαριστώ, Ντόρι. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα άκουσα ότι ο σταθμός αυτός έκλεισε μέσα σε λίγες ώρες και πραγματικά σοκαρίστηκα. Πιστεύω ότι παρότι σαφώς και είναι απαραίτητο να υπάρξει δημοσιονομική εξυγίνηση στην Ελλάδα γενικότερα και στο σταθμό κυρίως, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διεξήθησαν όλα αυτά είναι απαράδεκτος. Δεν έχουν καμία σχέση με συμμετοχική δημοκρατία, όπου καλείται κανείς να ε, τοποθετηθεί ε, για δύσκολα θέματα. Το να μην υπάρχει όμως σήμα να έχουμε μία μαύρη οθόνη, ε, αυτό είναι απαράδεικτο σε μία δημοκρατία, έστω και με κρίση. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι που αποφάνθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, που είπε ότι πρέπει πλέον να εκπέμπεται σήμα. Βέβαια η συζήτηση για τον αριθμό του προσωπικού και τον προσανατολισμό, αυτό θα ακολουθήσει και πρέπει να ακολουθήσει. Γιατί όπως είπε και η Ντόρις, τα κόμματα ε, τα τελευταία χρόνια τοποθέτησαν εκεί πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν ήταν προς όφελος του σταθμού. Ε, ούτε και αυτό είναι δυνατό να συνεχιστεί, ε, όμως οι εξελίξεις αυτές είναι μπούμεραγκ για αυτούς που αποφάσισαν. Φαίνεται ότι έτσι ήταν τα πράγματα στην Ελλάδα, έτσι γινόντουσαν. Κατόπιν τούτου καλούνται και όλοι να ασκήσουν αυτοκριτική, αλλά δεν είναι δυνατόν για καθαρά δημοκρατικούς λόγους να κλείνει ένας κρατικός ραδιοσταθμός. Ε, και θεωρώ ότι η απόφαση που έχει ληφθεί είναι σωστή. Πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό είναι και δική μας προτεραιότητα, να υπάρχουν εύρυθμα λειτουργούντες ε, κρατικοί στεθμοί. Απλά πρέπει να το εξασφαλίσουμε αυτό. Ο κύριος Μιγκάλσκι. Ο Μπόρις, προηγείται ο Μπόρις. Ευχαριστώ τον κύριο Μιγκάλσκι, που μου άφησε λίγα λεπτά. Θα ήθελα να πω ότι οι μέθοδοι που ακολουθήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση είναι αντιδημοκρατικές. Φυσικά ο τηλεοπτικός εκείνος σταθμός άπρεπε να έχει αναδιαρθρωθεί, ίσως να χρειάζονταν και απολύσει γιατί η οικονομία είναι ανελαίτη, αλλά από τη στιγμή που χάνεται το σήμα, δεν εκπέμπει καθόλου ο σταθμός και κλείνεται η κρατική ορχήστρα και όλος ο κόσμος βλέπει τους μουσικούς να κλαίνε. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Δηλαδή, δεν πρέπει να είναι πολιτική η τηλεόραση, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου εχθές που ακύρωσε την απόφαση του Πρωθυπουργού Σήμερα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα που να λέει ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιες μεθόδους. Πώς θα οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων εάν βλέπουμε την Τρόικα που ευθύνεται για την κατάσταση, όπως θεωρεί ο κόσμος τουλάχιστον, και απ' την άλλη να κλείνει η τηλεόραση και η κρατική ορχήστρα. Δεν γίνεται έτσι εμπιστοσύνη στους πολίτες. Κοιτάξτε, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες το θέμα ε, κατά πόσον μπορεί πράγματι να διατηρηθεί μια φιλαρμονική όχι. Κοιτάξτε, τώρα μην τον μπερδεύουμε αυτό, μην τον μπερδεύουμε με την, ε, ε, το πλήρως αντιδημοκρατικό κλείσιμο ενός σταθμού. Το να μην υπάρχει μια φιλαρμονική, αυτό μπορεί να φύλλεται σε δημοσιονομικούς λόγους. Μην τα μπερδεύουμε, γιατί μιλάμε για χώρες που μαστίζονται από την κρίση και κάπου πρέπει να βρίσκουμε, κάπου πρέπει να πούμε τα λεφτά. Μην μπερδεύουμε τώρα ε, τα μήλα με τα πορτοκάλια. Ε, τώρα, κατά πόσο ήσαν σωστό ή λάθος δεν το ξέρω αυτό, αλλά για άλλα πράγματα μιλάμε. Ο κύριος Μιγκάλης και έχει το λόγο. Να Ζήτησα να δοθεί ο λόγο του κ. Μπόρης. Πρώτα, αλλά εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Ήδη πολλές φορές έχουμε μιλήσει για τα δημόσια μέσα μαζικής ενημέρωση, τα οποία είναι απαραίτητα για την δημοκρατία σήμερα. Ουσιαστικά οικοδομούν ε, κάτι που δεν ε, οικοδομείται από τα ιδιωτικά μέσα πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό που έγινε στην Ελλάδα. Το παράδειγμα της αντίδρασης του ελληνικού δικαστηρίου δείχνει ότι οι Έλληνες τα καταφέρνουν από μόνοι τους τελικά και πρέπει να σκεφτούμε μήπως ε, δεν είναι απαραίτητη τελικά μια παρέμβαση από τις Βρυξέλλες. Ε, οι Έλληνες μπορούν να τα καταφέρουν πολύ καλά και μόνοι τους. Όμως φυσικά και εγώ λυπάμαι για το κλείσιμο της ΕΡΤ, αλλά από τη μία λέμε στους Έλληνες να κάνουν δραστικές εξοικονομήσεις, δραστική οικονομία και τη στιγμή που κάνουν κάτι τέτοιο, παραδείγματο χάρη, ε, στην περίπτωση αυτή ανησυχούμε. Έτσι λοιπόν έχω μια αμφιβολία εδώ. Μήπως ε, επιδεινώσουμε την κατάσταση αν παρέμβουμε και μήπως αυτή η επιφυλακτικότητα που υπάρχει απέναντι στις Βρυξέλλες ε, θα αυξηθεί. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να λαμβάνω υπόψη στην Ελλάδα. Η Πέτρα. Η Πέτρα, ε, θέλω να πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα και ε, να μην ξεχνάμε το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ, όπου είπαμε με απόλυτη σαφήνεια ότι βεβαίως η οργάνωση των μέσων ενημέρωσης ε, είναι θέμα των κρατών μελών. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι είναι καθήκον του Κοινοβουλίου σε μια τέτοια κατάσταση να πει με απόλυτη σαφήνεια ότι ε, ορισμένες συμπεριφορές κάτω από το πρίσμα της δημοκρατίας είναι απαράδεκτες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα αναμειχθούμε στο πώς θα διαμορφώσουν στο μέλλον την κρατική τηλεόραση, να πούμε μόνο ότι ελπίζουμε να βρουν ένα δρόμο, μια λύση ε, η τηλεόραση ε, στο μέλλον να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του ελληνικού λαού. Για να κλείσουμε λοιπόν, το ε, δικαστήριο είπε ο σταθμός να εκπέμπει σήμα, να λειτουργεί. Και διαβάζω το εξής. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε συμβιβαστική λύση με βάση την οποία ε, η ΕΡΤ θα αρχίσει να εκπέμπει σήμα. Ε, μία τριμερής ε, διακομματική επιτροπή προσωρινά θα προσλάβει κάποιους δημοσιογράφους και έτσι θα λειτουργεί η τηλεόραση μέχρι να θεσπιστεί σχετική νομοθεσία για τον κρατικό ε, σταθμό. Ο Πρωθυπουργό ε, συμφώνησε ε, και είπε μάλλον ότι θα πρέπει να συρρυκνωθεί. Άρα δηλαδή αυτός να βγάλει τους δικούς του, αυτούς που έβαλε εκεί και οι άλλοι να βγάλουν και εκείνοι τους δικούς τους. Δυστυχώς έτσι γινόντουσαν τα πράγματα στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι ανακατευόμαστε και επεμβαίνουμε, αλλά όταν σε ένα ευρωπαϊκό κράτος ξαφνικά κλείνει ένας ε, κρατικός σταθμός, αυτό μας ε, αγγίζει. Ε, βέβαια, από ό,τι φαίνεται, οι Έλληνες δεν φλέγονται και μου λέγανε σε να μιλήσουμε, να μιλήσουμε. Το κάναμε και νομίζω ότι τελικά, τέλος πάντων, εμείς μεταξύ μας όλοι συμφωνούμε. Η κυρία Βερζιά ζήτησε συγγνώμη, είπε ότι δεν μπορεί να παρίσταται, έστειλε μία επιστολή στους συντονιστές. Νομίζω το θέμα έχει κλείσει γιατί αποφάσισε το δικαστήριο, συμμορφώθηκε η κυβέρνηση, τέλειωσε το θέμα. Τι να πούμε άλλο. Εμείς δεν είμαστε για να λύσουμε τα προβλήματα της Ελλάδας. Προφανώς αυτά είναι θέματα των Ελλήνων. Αλλά δεν έπρεπε να το κάνουν αυτό που έκαναν και γι' αυτό συζητήσαμε το θέμα. Κλείνει λοιπόν και νομίζω ότι θα παρακολουθούμε την κατάσταση, αλλά είμαι σίγουρος ότι ε, θα βρούνε μια λύση που δεν θα σημαίνει όμως 2,5 ή 2.650 πάλι γιατί αυτό δεν γίνεται. Πάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης. Ε, The editorial director of information programming of Belgium. Πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων με τους κυρίους Αλιαξέη Τζίκα Τιβίσκη, της Μπελζάτ, τη Ρατζίνα, ε, Ναταλία Ρατζίνα και τον ε, κύριο Γουάπα από το Ράντιο Ράσια. Πρόκειται, η τελευταία κυρίως είναι μια ανεξάρτητη, ε, ένας ανεξάρτητος σταθμός στη Λευκορωσία. Έχουμε μία μετάφραση στα ρωσικά μάλλον διερμηνείς ε, Ρώ, Ρώσους. Ποιος θέλει παρακαλώ να ξεκινήσει. Η Νατάλια Ρατζίνα έχει το λόγο. Yes, uh, thank you for the invitation. I will speak Russian if it's possible. ευχαριστώ για την πρόσκληση. είναι δυνατόν θα μιλήσω ρωσικά. Έχω πάρα πολλά να σας πω, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. χάρτη 97 είναι ε, το πιο δημοφιλές, ε, δημοφιλές ε, νέων στη Λευκορωσία και το 2010, από το 2010 το καθεστώς Λούκοσενκο ε, που ουσιαστικά κατήργησε την ανεξάρτητη τηλεόραση έκανε ακόμη μεγαλύτερα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση σκοτώθηκε ο κ. Παπενίν ε, τρεις ε, ποινικές έρευνες ξεκίνησαν και δύο φορές μας κατάσχεσαν τον εξοπλισμό στις 19 ε, Δεκεμβρίου 2012 αστυνομικοί έκαναν ε, έφοδο στα γραφεία μας και εμένα με φυλάκισαν και με κατηγόρησαν για Ε, ανώφευση των ε, εκλογικών αποτελεσμάτων. Εγώ έπρεπε λοιπόν να διαφύγω από την ε, Λευκορωσία και αυτό το έκανα γιατί ήθελα να είμαι αμερόληπτη δημοσιογράφος. Οι αμερόληπτοι και ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι σήμερα δεν μπορούν να δουλέψουν στη Λευκορωσία γιατί δέχονται συνεχείς πιέσεις από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Και αυτή η πίεση ασκείται σχεδόν ε, καθημερινά. Επίσης, ε, προσπάθησα να διαφύγω από τον έλεγχο τη ΚΑΓΚΕΜΠΕ, την οποία μπορούσα να ελεγχθώ εκεί, μπορούσα να νιώσω εκεί. Σήμερα ε, εκπέμπουμε από την Πολωνία και είναι και μια χώρα όπου και η Μπελσάτ και η Ράτια εκπέμπουν και λειτουργούν μπορούμε να εργαστούμε στην ε, Πολωνία και έχουμε πάνω από 100.000 επισκέπτες την ημέρα. Η πολωνική κυβέρνηση μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, όμως δεν αρκεί, γιατί υπάρχει έλλειψη πόρων. Και ξέρουμε ότι οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να ασκήσουν το επάγγελμα τους ε, με πολλή υποστήριξη ε, κατά τις ε, προεδρικές εκλογές του Παμά και είναι πολύ σημαντικό σήμερα λοιπόν να υποστηρίξετε τα ανεξάρτητα μέσα της Λευκορωσίας ε, δεν είναι και τόσο πολλά. Μιλάμε για τα δική μας ιστοσελίδα και το ραδιόφωνο ράντια προκειμένου να διασφαλίσουμε την η πληροφόρηση φτάνει στους πολίτες μας. Επίσης, ε, δεν θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας και εντό Λευκορωσίας ε, και να αναπτυχθούμε και στο τομέα του εντύπου. Χρειαζόμαστε πολύ συγκεκριμένη υποστήριξη. Η χρηματοδότηση που λάβουμε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που λαμβάνουμε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν επαρκεί ή ίσως δεν χρησιμοποιείται ορθά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρετε ότι δέχεται ε, να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι του Στάλιν ε, στη Λευκορωσία. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Εγώ μπορώ να το βεβαιώσω αυτό ως πρώην πολιτική κρατούμενος. Χρειαζόμαστε λοιπόν αλληλεγγύη και σαφή στρατηγική απέναντι στη Λευκορωσία. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία τέτοια στρατηγική. Ακούμε διάφορες δηλώσεις ε, και μπορούμε να δούμε ότι και η χρηματοδότηση που έχει ενεργοποιηθεί για τη Λευκορωσία δεν χρησιμοποιείται αποτελεσματικά. Ο Λουκασέγκο σκοτώνει χιλιάδε ανθρώπους, όμω, ε, η ζωή αυτών των πολιτών δεν είναι μόνο στα χέρια του Λουκασέγκο, αλλά και στα δικά σας χέρια, γιατί μπορείτε πράγματι να μα βοηθήσετε. Ευχαριστώ. Και εμεί σα ε, ευχαριστούμε. Οι ερωτήσει θα τεθούν ε, αργότερα. Παρακαλώ, ε, επόμενος ο μιλητής, ε, σας παρακαλώ ποιος ε, θα λάβει το λόγο. Λέγομαι Αλεξέη Τζουκάκη Βίτκη. Κύριοι Ευρωβουλευτέ, συνάδελφοι, λέγομαι Άλεξ Τζικαβίτσκι και εκπροσωπώ εδώ το μόνο ανεξάρτητο τηλεοπτικό σταθμό τη Λευκορωσία μέσω Ιντερνετ και δορυφόρου. Καταρχήν ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα τον Ευρωβουλευτή Μιγκάλσκι για την πρόσκληση. Άρχισα μιλώντας αγγλικά, αλλά ε, διότι ακόμη κι αν η Πολωνία δεν είναι το πλουσιότερο μέλος της Ένωσης, αποφάσισε να μας υποστηρίξει και να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας ε, ανεξάρτητης τηλεόρασης χωρίς διοργοκρισία. Μερικοί θεωρούν ότι αυτό είναι αδύνατον, αλλά για να αποτύσσω να φόρο τιμή στην Πολωνία θα συνεχίσω στα παλωνικά. που πολύ συχνά υπήρξαν φυλακίσεις των δημοσιογράφων που ποτέ όμως δεν υπέκυψαν. Εδώ και πέντε χρόνια συνεχίζουμε να εκπέμπουμε πλήρες πρόγραμμα δυστυχώς από τη Βαρσοβία. Γιατί από τη Βαρσοβία και γιατί δυστυχώς, διότι όταν εργάζεται κανείς σε μία χώρα θα εκπέμπει προς μία χώρα, θα ήθελε να εργάζεται και σε αυτήν. Στη Λευκορωσία όμως, στη χώρα μου δηλαδή, υπάρχει μια δικτατορία που δεν ανέχεται την ελευθερία της έκφρασης και της σκέψης. Δεν επιτρέπεται ανεξάρτητη τηλεόραση και ραδιόφωνο. Μαζέψαμε λοιπόν μια ομάδα θαραλέων δημοσιογράφων και εκπέμπουμε από την Πολωνία. Γιατί στην Πολωνία θυμούνται ακόμη τι ήταν η κομμουνιστική φυλακή. Θέλησαμε να ανοίξουμε ένα γραφείο στη Λευκορωσία και αυτό το απαγόρευσαν. Και στον Πιάλιστο, στα σύνορα με την Πολωνία, υπάρχουν τα γραφεία της Χάρτας 70 που εκπέμπει από το Ιντερνετ. Η Πολωνία λοιπόν μας βοήθησε Καταφέραμε επίσης να εκπέμψουμε και μέσω δορυφόρου ώστε οι Λευκορώσοι να μπορούν να μας βλέπουν. Οι τηλεθεατές μας και οι ακροατές μας αυξάνονται συνεχώς. 895.000 θεατές έχουμε, τηλεθεατές, πάνω από 12% δηλαδή του ενήλικου πληθυσμού. 39% των κατοίκων της Λευκορωσίας γνωρίζουν την ύπαρξή μας και έχουμε και την υποστήριξη του 77% των τηλεθεατών γενικότερα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 17 ώρες προγράμματος την ημέρα χρησιμοποιούμε περίπου 200 εργαζόμενους στη Λευκορωσία, την Πολωνία και τη Λιθουανία. Όπως ξέρετε βέβαια είναι πολύ ακριβή η λειτουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού και ευχαριστούμε την πολωνική κυβέρνηση που μας χρηματοδοτεί αλλά και την υπηρεσία SDA της Φρουητίας καθώς και την Ορβηγία και το Συμβούλιο Βορείων Υπουργών και το Ολλανδικό Σχέδιο Μάτρα. Μην ξεχνάτε ότι όταν βοηθάτε εμάς βοηθάτε όχι μόνο τη δική μας τηλεόραση και ραδιόφωνο αλλά και την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων μην ξεχνάτε ότι η Λευκορωσία ήταν χώρα ευρωπαϊκών παραδόσεων που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακριβώς στα σύνορα με την Ένωση. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στη Λευκορωσία χάρη στις εκπομπές μας. Πολλές ελπίδες έχετε, αισιόδοξοι είστε. Ο Ευγένιος Βάπας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, εκπροσωπούμε μέσα μαζικής ενημέρωσης που αντιτίθενται στο μονοπόλιο του Αλεξάνδρου Λουκάσινκου. Είναι ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και Πόσες φορές ζητήσαμε αναγνώριση επίσημη από το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών και άλλων χωρών μας τα απέρριψαν. Δεν υπάρχει λοιπόν ομαλοποίηση της κατάστασης στην Λευκορωσία αλλά συνεχίζεται η καταπολέμηση της ανεξάρτητης ενημέρωσης. Τα τρία μέσα που εκπροσωπούνται εδώ είναι σημαντικές πολιτιστικές αιστείες για την Λευκορωσία γιατί ένας ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός δεν είναι μεν καθεαυτό κάτι που είναι από μόνο του μόνο σημαντικό αλλά εκπροσωπεί και ολόκληρο κοινωνικό κίνημα. Ο Λουκάσενκο θέλει να διαιρέσει το λαό ενώ με μας μπορούν να εκφραστούν και οι Λευκορώσοι. Εκτός του μονοπωλίου ο Λουκάσενκο θέλει να καταπολεμήσει τον πολιτισμό στο σύνολό του. Εδώ στη συνεδρίαση της Επιτροπής σας θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι πολιτιστικές αιστείες καταπιέζονται και διώκονται στη Λευκορωσία. Και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε νομίζω να μας υποστηρίξει και να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και να αναπτυχθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη ένα γενικότερο όραμα. Και αυτό είναι δυνατόν μέσω των ανεξαρτήτων μέσων που εκπροσωπούμε. Δε, συχνά υποτιμούμε την πτυχή αυτή, αλλά από εκεί θα ξεκινήσει μια αλληλεγγύη μεταξύ όλων των Λευκορώσων. Εμείς οι Λευκορώσοι πρέπει να αυτοβοηθηθούμε καταρχάς. Αλλιώς χωρίς αυτό δεν θα είχαμε φτάσει μέχρι εκεί που φτάσαμε. Εναντίον μας βλέπουμε να υψώνονται όλα τα μέσα ενός κράτους και εμείς έχουμε ένα πατίνι απλώς για να το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό σημαίνει ότι φυστάμεθα και επιθέσεις, hacking δηλαδή και άλλα τέτοια μέσα που χρησιμοποιεί ο Λουκάσενκο για να μπλοκάρει τις εκπομπές μας γιατί ξέρει ότι αν πετύχει, αν αποτύχει μάλλον αυτή η παρεμπόδιση, τότε η λευκορωσική κοινωνία θα έχει τελικά πρόσβαση σε ελεύθερη πληροφόρηση. η πολωνική κυβέρνηση είναι υποδειγματική στην υποστήριξή μας και έτσι μπορείτε και εσείς να τα μαθαίνετε όλα αυτά. Έχουμε ετοιμάσει μπροσούρες στα αγγλικά. Θα σας τις μοιράσουμε. Μην ξεχνάτε ότι οι δημοσιογράφοι είναι μέρος του πολιτισμού. Μην επιδείξετε λοιπόν αδιαφορία ή ουδετερότητα. Τέλεια. Ε, Πρόεδρος, όπως ξέρουμε, η ε, από τη Λευκορωσία παρουσιάσατε την κατάσταση ως πάρα πολύ δυσάρρωστη. Ε, στη θέση 150 βρίσκεται η Λευκορωσία όσον αφορά την ελευθερία του τύπου, που είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Και όσον αφορά τις ε, δημοκρατικές διαδικασίες, οι δημοκρατικές διαδικασίες μπορούν να επικρατήσουν σε μια χώρα μόνο εφόσον η δημοκρατία στηρίζεται από τα μέσα ενημέρωσης. Μόνο δηλαδή εφόσον οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε όλες τις αξίες ε, της δημοκρατίας. Η Χέλγα έχει το λόγο και μετά ο Λόταρ. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους τρεις σας ε, θερμά για τις ε, πολύ ξεκάθαρες απόψεις που εκφράσατε. Καταστήσατε απόλυτα σαφές πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη για την προβολή της υπόθεσης ε, που θέλετε να προβάλλετε. Μιλάμε για δυστυχώς μια δικτατορία που υπάρχει στη Λευκορωσία και με δύναμη και αποφασιστικότητα και κατηγορηματικότητα μας καταδείξατε πόσο σημαντική είναι η δουλειά σας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μας δείξατε το ότι Λόγω του πολιτισμού σας ε, θα θέλατε κι εσείς να νίκετε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Αυτά πραγματικά εμείς πρέπει να τα στηρίξουμε. Και χαίρομαι που μας δόθηκε σήμερα η ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας. Είναι απαραίτητο πράγματι στη χώρα σας ε, να υπάρξει ε, κοινωνία των πολιτών. Είναι σημαντικό να μας ενημερώνετε για αυτές τις προσπάθειες. Αυτά που ακούσαμε σήμερα ήταν μια πολύ σημαντική συνδρομή χώρα Εσείς ε, σήμερα μιλήσατε για το θέμα της ε, στρατηγικής της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατά την άποψή σας η στρατηγική αυτή δεν είναι επαρκώς διαυγής. Ε, ίσως μπορείτε σύντομα να μας πείτε λιγάκι κατά την άποψή σας τι πρέπει ακόμα να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο κατηγορηματική στην στρατηγική της προσέγγισης απέναντι στη Λευκορωσία. Ο κύριος Λούτα Μπίσκι. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Η Λευκορωσία παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα. Συμπτωματικά ε, στο Πότσταμ που ήμουνα, ε, το Πότσταμ έχει αδελφοποιηθεί με το Μίνσκ. Ε, και Γι' αυτό έχω πάει ε, πολύ συχνά στο Μίνσκ και έχουμε και πολύ καλούς φίλους από το Μίνσκ που μας ε, επισκέφτηκαν. Ξέρω λοιπόν ότι ζείτε κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες ε, συνθήκες. Ξέρω ότι η δουλειά σας ως ελεύθερη δημοσιογράφη είναι σχεδόν αδύνατη στη Λευκορωσία. Άρα δηλαδή πρέπει απαραίτητα να σας στηρίξουμε ηθικά τουλάχιστον, όχι οικονομικά, να στηρίξουμε εσάς και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εσείς ε, πραγματικά ενσαρκώνετε το, την προσπάθεια η Λευκορωσία στο μέλλον να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας εύχομαι λοιπόν κουράγιο στην προσπάθειά σας αυτή. Ευχαριστούμε Λούτα. Ε, ο Πιότρ έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μάρκ Γκαλσκή για την πρωτοβουλία αυτή Λυπάμαι που εδώ έχουμε πόντες ε, σήμερα, γιατί η Ευρωπή είναι... Μπορούμε να τη δούμε και από γεωγραφική σκοπιά, δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν ε, βλέπουμε ότι λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορά μας έχουμε να κάνουμε με την τελευταία δικτατορία αυτού του ιστορικού τμήματος της Ευρώπης ε, και δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να υποστηρίξουμε αυτή τη χώρα. Πέρα από την πολιτική υποστήριξη, που είναι πολύ σημαντική σήμερα, είναι πολύ σημαντικό και το θέμα της πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης, γιατί μιλάμε για την πρόσβαση στην αλήθεια. Έτσι λοιπόν, σήμερα στην Λευκορωσία έχουμε ε, το φόβο να βασιλεύει. Όμως ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε το 90% των πολιτών της Λευκορωσίας που ποτέ δεν έχουν βγει από τα σύνορα, δεν έχουν ε, περάσει τα σύνορα για να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε λοιπόν πώς έχουμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην πληροφόρηση. Ευχαριστώ όλες τις κυβερνήσεις και όλες τις χώρες που υποστηρίζουν οικονομικά το εγχείρημα, αλλά ήθελα να ζητήσω και από μας και από τη δική μας Επιτροπή να ενεργοποιήσει κάποια μέσα, κάποια κονδύλια που υπάρχουν στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής σχέσης, ανατολικής εταιρικής σχέσης, για να βοηθήσουμε τα ανεξάρτητα μέσα. Υπάρχουν τα τεχνικά μέσα. Αυτό που λείπει είναι η χρηματοοικονομική υποστήριξη. Και ξέρω ότι υπάρχουν κάποια κονδύλια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της εταιρική σχέσης. Και θα πρέπει να βρούμε μια γραμμή στον προϋπολογισμό που προτείνουμε. για αυτή την πολιτική γετνίασης και με σχέσης με την Ανατολή. Ευχαριστώ. Κύριος Μικάλσκι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Προεδρείο της Επιτροπής μας, γιατί χάρη σε αυτούς μπορέσαμε να οργανώσουμε αυτή τη συνάντηση. Και να Έχουμε εδώ την παρουσία τριών σημαντικών μέσων, μια ιστοσελίδα ενό καναλιού και ενό ραδιοφώνου. Πράγματι, γειτονεύουμε με ένα δικτάτορα. Είναι ακριβώς στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο δικτάτορας αυτός. Βρίσκεται ακριβώς στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δολοφονεί τους ανθρώπους, τους φυλακίζει και εμείς τον δεχόμαστε ως γείτονα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Πιότρ ότι υπάρχουν τα μέσα Υπόθηκε ότι ίσως μπορούμε να υποστηρίξουμε και ηθικά τη Λευκορωσία, όμως πολιτική και ηθική στήριξη υπάρχει αρκετή εδώ και καιρό. Αλλά αυτό που χρειάζεται τώρα είναι οι επενδύσεις ε, στα μέσα. Αν δεν, υπάρξει, αν δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην ενημέρωση και στην ανταλλαγή απόψεων, αν ε, δεν υπάρχει πρόσβαση των Λευκορώσων που ζουν σε ένα κλειστό κύκλο, Δίχως όλα αυτά δεν θα αλλάξουν οι συνειδήσεις και η δικτατορία του Λουκασέγκο θα υποστηρίζεται μέσω της άγνοιας των πολιτών. Πρέπει λοιπόν να παράσχουμε συγκεκριμένη υποστήριξη φυσικά. Αυτή η συγκεκριμένη υποστήριξη σημαίνει τη χρηματοοικονομική υποστήριξη και ο κύριος Μπορίς ε, το είπε ήδη, τα χρήματα υπάρχουν. Ε, swoje problemy na forum unijnym. Όμως ε, σήμερα ε, το ότι έχουμε τρεις ε, εκπροσώπους εδώ των μέσων που μπορούσαν να παρουσιάσουν τα προβλήματα που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα βήμα προς ε, την ενημέρωση των πολιτών. Και ευχαριστώ λοιπόν ε, την Προεδρία αυτής της Επιτροπής. Κοιτάξτε, θέλω να υπογραμμίσω ότι προφανώς ε, και παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά τι διαδραματίζεται ή τι δεν γίνεται στη Λευκορωσία. Ε, και στην Επιτροπή μας συζητήσαμε για την εκδήλωση αυτή του ice hockey στη Λευκορωσία και είπαμε μα πώς είναι δυνατόν να γίνεται εκεί αυτή η εκδήλωση όπου οι άνθρωποι ποδοπατούνται και τα δικαιώματα πόσο μάλλον και οι θύνοντες εκμεταλλεύονται αυτήν την ε, οργάνωση, την εκδήλωση απλά και μόνο για να προβληθούν. Ε, γράψαμε λοιπόν στην Ένωση, στην Ομοσπονδία του Hockey επιπάγου να το σκεφτούν το κατά πόσον θα πρέπει να οργανώνουν ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε μια χώρα όπου δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γνωρίζετε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς και άλλοι ανησυχούν πάρα πολύ ως προς την ε, διαβίωση ε, τα δικαιώματα των πολιτικών κρατουμένων. Ε, προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Εντάξει, κάποιοι είναι πιο επώνυμοι από άλλους, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, όλοι υποφέρουν. Το θέμα ε, ότι απλώς ε, στυλιτεύουμε ορισμένα πράγματα θα πρέπει κάποτε να αποδώσει κιόλας. Αλλά βέβαια στις δικτατορίες δυστυχώς προσκρούει κανείς πάντα σε μη ακούοντα ότα. Είπατε ότι τα χρήματα δεν επαρκούν και είπατε και ότι τα κονδύλια, τα χρήματα δεν διοχετεύονται σε σωστούς σκοπούς. Και ρωτώ, τι χρήματα παίρνετε, από ποια γραμμή, από ποιο κονδύλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πού παίρνετε τα λεφτά σας, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, τι είδους αποδείξει αποδείξεις υπάρχουν. Μπορείτε λιγάκι να μας ε, αποδείξετε γιατί ε, διοχετεύονται λανθασμένα τα χρήματα αυτά. Έτσι ώστε εμείς ως βουλευτές να πούμε στην Επιτροπή προσέξτε όταν δίδετε χρήματα στη Λευκορωσία αυτά χάνονται κάπου, δεν φτάνουν εν πάση περιπτώσει ε, στο σκοπό τους. Ναι, θα προσπαθήσω να απαντήσω την ερώτησή σας και την ερώτησή σας σχετικά με τη στρατηγική. Όμως ε, θα πρέπει να φύγω σύντομα γιατί έχω μια συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, η ευρύτερη υποστήριξη γίνεται τώρα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας. Δυστυχώς, οι πόροι αυτοί δεν αρκούν. Μας επιτρέπουν να λειτουργήσουμε για έξι μήνες περίπου, όχι περισσότερο επίσης. Λαμβάνουμε μια μικρή χρηματοδότηση από το Ταμείο Μάρσελ, από τη Γερμανία και από την Ορβηγία. Και πέρσι Λάβαμε υποστήριξη από το Ταμείο Μάτρα, από τις κατοχώρες, όμως δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε αύριο να εκπέψουμε, να λειτουργήσουμε, γιατί η υποστήριξη είναι πολύ μικρή και ακολουθείται μια προσέγγιση Υποστήριξη ένα τεμάχιο. Ε, θέλουμε υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως υπάρχει τόσο μεγάλη γραφειοκρατία που φοβούμαστε για το μέλλον, ε, γιατί εγώ για να διαχειριστώ ε, όλη αυτή τη γραφειοκρατία και να δώσω τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να προσλάβω περισσότερους ανθρώπους από τους δημοσιογράφους και αυτό δεν είναι βιώσιμο γιατί το θα πρέπει να πληρωθούν και οι άνθρωποι αυτοί. Ε, και αν πληρώσουμε τους ανθρώπους που θα δεκπαιρεώσουν τα έγγραφα, τότε δεν θα έχουμε αρκετά χρήματα για δημοσιογράφους. Χρειαζόμαστε λοιπόν απλουστευμένες διαδικασίες. Νομίζω ότι μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. γιατί νομίζω ότι μπορείτε να μας δώσετε υποστήριξη έτσι όπως δόθηκε υποστήριξη στο, εργα... στο Συνδικάτο Αλληλεγγύης στην Πολωνία. Λοιπόν, Τώρα, δεν ε, θα έπρεπε να έρθουν οι κυρώσεις ε, κατά του καθεστώτος Λουκασένκο, γιατί η κατάσταση ολένα και επιδεινώνεται. Οι μυστικές υπηρεσίες ελέγχουν τα πάντα στη χώρα και γι' αυτό υπάρχουν κάποιοι ευρωβουλευτές όπως ο κύριος ε, Λέσκη που κατέληξε σε συμπέρασμα ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση, όμως η αλήθεια είναι ότι πολλοί πολιτικοί ακτιβιστές έπρεπε να διαφύγουν από τη χώρα. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να ενδυναμωθούν οι κυρώσεις κατά του καθεστώτος. Επίσης, είναι απαραίτητο να εισαχθούν, να επιβληθούν κυρώσεις κατά των επιχειρηματών που χρηματοδοτούν το καθεστώς Λουκασένκο και πρέπει να εισαχθούν για κάποιες χειρουργικές ε, κυρώσεις, παραδείγματο χάρη σε ό,τι αφορά το εμπόριο σε πετρελαϊκά προϊόντα, γιατί και τα έσοδα από αυτό το εμπόριο πάνε κατευθείαν ε, στη χρηματοδότηση των μυστικών υπηρεσιών που βασανίζουν και δολοφονούν τους πολίτες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε υποστήριξη. Πρέπει να υποστηρίξετε τις οργανώσεις και τους ακτιβιστές ανθρωπινών δικαιωμάτων και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει διευκόλυνση του καθεστώτος θεωρήσεων ε, για τους ε, πολίτες για να μπορούν ε, να επισκεφθούν την Ευρώπη και θα πρέπει να δίνονται και δωρεάν οι θεωρήσεις για τους ανθρώπους αυτούς. Αυτό θα αλλάζει ριζικά την κατάσταση. Είδαμε ότι το καθεστώς Λουκασένκο υπάρχει εδώ και 20 χρόνια και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Αν τίποτα όμως δεν αλλάξει και στο μέλλον θα κρατήσει 20 χρόνια ακόμα. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα της ε, Λευκορωσίας, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να μιλήσουμε και για τη Ρωσία, γιατί αν δεν υπήρχε η Ρωσία δεν θα μπορούσε να σταθεί το καθεστώς. Η Ρωσία είναι σημαντικός εταίρος για τη Λευκορωσία. Εντάξει, ε, μπορείτε να κάνετε συναλλαγές με τη Ρωσία, αλλά θα πρέπει να μιλάτε μαζί τους και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς ε, στο Μπενσάτ ε, όταν έχουμε προσκεκλημένους ε, μας θέτουν ερωτήσεις για τον προπολογισμό. Λέμε ότι μιλάμε για 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και όταν τους λέμε αυτό ξεσπούν στα γέλια, νομίζουν ότι τους κοροϊδεύουμε. 6 εκατομμύρια ε, είναι για ένα μήνα, ρωτάνε. Αυτή είναι η πολωνική υποστήριξη. Υπάρχουν βέβαια και μικρές επιδοτήσεις ε, που έρχονται να συμπληρώσουν τη χρηματοδότησή μας. Όμως ε, τα μέσα μας δεν αναπτύσσονται, δεν προσελκύουν νέα, νέους θεατές. Το κρατηριό μας είναι σε τέλμα. Για να αναπτυχθούμε χρειαζόμαστε και 2-3 εκατομμύρια από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλά, όχι δεν νομίζω. Αυτή τη στιγμή δεν παίρνουμε ούτε ένα ευρώ απευθεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, το ραδιοφωνό μα ε, να σας πω ότι υπάρχει από το 1988 και το 2006 ανανεώσαμε ε, το σήμα ε, εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο σε περιοχές ε, όπου έχουμε μισό εκατομμύριο λευκορώσους. Ε, το πολωνικό κράτος χρηματοδοτεί 100% τη λειτουργία μας. Έχουμε 62 υπαλλήλου. Φυσικά βοηθούν και κάποιε άλλε χώρε, Αυστρία, κάτω χώρε, Ηνωμένο Βασίλειο, κάποια ιδρύματα, ανεξάρτητα. αν ε, μπορούμε να εκπέμπουμε 24 στο 24 ώρο με ένα προπολογισμό ενό εκατομμυρίου το χρόνο, βλέπετε ότι βλέπουμε πώς θα ξοδέψουμε και το κάθε ευρώ. Εμείς ε, για να μπούμε σε πραγματικό ανταγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουμε τόσο ισχυρά μηχανήματα όπως ε, και οι αντίπαλοι μας πίσω από τα σύνορα. Στη Λευκορωσία υπάρχουν 24 ε, ραδιοφωνικοί σταθμοί στα FM που χρηματοδοτούνται από το καθεστώς. Θέλουμε εμείς να είμαστε σοβαροί, όμως είναι πάρα πολύ μεγάλες οι προκλήσεις. Ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα θαύμα. και να μην κάνουμε τίποτα, πρέπει να αναλάβουμε δράση. Κοιτάξτε, μιλήσατε προηγουμένως για θέμητο ανταγωνισμό. Αυτό μάλλον αστείο είναι, γιατί η κατάσταση είναι θλιβερή. Είσαστε σε μια κατάσταση όπου είσαστε αποκλεισμένοι, δεν μπορείτε καν να ανταγωνιστείτε. Είσαστε εκτός και εξαρτάστε από βοήθεια από όπου και να έρχεται αυτή, από ιδρύματα, από κυβερνήσεις, ε, ε, από τους Πολωνούς που μπράβο τους. Ε, το θέμα είναι, είπατε ότι παίρνετε 200.000 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα χρήματα σας δίδονται εύκολα ή μήπως σας αναγκάζουν να συμπληρώνετε έντυπα επί εντύπων, γιατί η συνάδελφό σας προηγουμένως ε, είπε ότι αν θέλει κανείς να πάρει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει καταρχήν να έχει προσλάβει πάρα πολλούς υπαλλήλου για να χρηματοδοτηθεί. Ε, σε εσά τι συμβαίνει, μπορείτε εύκολα να πάρετε τις 200.000. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε, γιατί όταν θα απευθυνθούμε σε άλλους υψηλότερα ιστάμενους πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα προβλήματα. Κοιτάξτε, η κατάσταση έχει ως εξή. Πρέπει να προσλάβουμε κάποιον, να προσλαμβάνουμε ανθρώπους που 100% να είναι αφοσιωμένος στην παρακολούθηση των ευρωπαϊκών διαγωνισμών και των εμπειρογνωμών. Δεν έχουμε όμως τη δυνατότητα, μας αρνήθηκαν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις γιατί οι ενωσιακές αρχές μας βαθμολόγησαν με 19,6 στα 20 που ήταν λέει η βάση για να προχωρήσουμε και ως εξήγηση της άρνησης αυτής του 0 2,4% μας είπαν ότι δεν έχουμε αρκετή τοπική εμπειρία στη Λευκορωσία, ενώ εμείς είμαστε εκείνοι που έχουν αυτή την εμπειρία. Και υποφελήθηκαν άλλοι από αυτά τα κονδύλια. Εμείς εκπέμπουμε 18-19 ώρες τη μέρα προς τη Λευκορωσία. Πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί κάτι ειδικά για τη Λευκορωσία για να μην αναγκαζόμαστε να συμπληρώνουμε όλα αυτά τα χαρτιά κάθε μέρα. Εύκολα βλέπει κανείς πώς λειτουργεί η τηλεόραση. Ανοίγει κανείς το κουτί και βλέπει αν υπάρχει το σήμα. Αλλά δεν μπορεί να δει αν τα χρήματα έχουν δαπανηθεί σωστά. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί κάτι για να επωφεληθούν και τα σημαντικότερα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τζικαβίτσκι γιατί εδώ και χρόνια γίνεται λόγος για υποστήριξη των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία. Η χάρτα, η τηλεόραση πρέπει, είναι αναγκασμένες να υποβάλουν συνεχώς αιτήσει για επιχορήγηση και δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιες άμεσες τις υποβολές αιτήσεων χρηματοδότησης. Αυτό είναι που ζητάμε και ζητάμε να, αλλαγεί, να αλλαχτεί. Να υπάρχει δυνατότητα στήριξης των λευκορωσικών ανεξάρτητων μέσων για να έχουμε τις επιχορηγήσεις άμεσα και να μπορεί να ακούγεται το ραδιόφωνο, ράτσια ή τηλεόραση και εδώ και παντού. Ζητούμε λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος, μια διαδικασία απλούστερη και πιο διαφανής γιατί αυτοί που επιχορηγούνται αυτή τη στιγμή είναι η, Λευ... η γραφειοκρατία της Λευκορωσίας. Τα πραγματικά ανεξάρτητα μέσα αποκλείονται. Κυρία Πρόεδρε, είδατε λοιπόν ε, τι γίνεται όταν έχουμε υπερβολικές ε, ρυθμίσεις. Το έχουμε ακούσει και σε άλλες περιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να προτείνω το εξής. Μήπως θα είχε νόημα οι δύο ε, συνάδελφοι που είπαν σχεδόν ε, τα ίδια ε, για τα κονδύλια να καταθέσουν μία γραπτή πρόταση που να την διαβάσετε εσείς περαιτέρω ως πρόεδρος ε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί τουλάχιστον αυτό το πρόβλημα δηλαδή να μην αυξηθεί το γραφειοκρατικό άχθος από τη χρήση των κονδυλίων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με πολύ σημαντική δουλειά θα ήταν λοιπόν ένα πολύ καλό παράδειγμα να συμβάλλουμε σε κάτι θετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Μπόρις έχει το λόγο. Θα ήθελα να... Θα είμαι σύντομος. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι σήμερα έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την υποστήριξη ενός ελεύθερου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού. Ε, τώρα αυτό στηρίζεται από την πολωνική κυβέρνηση. Πρέπει όμως να προχωρήσουμε πιο πολύ. Είμαστε μπροστά στην έγκριση ενός ε, νέου προϋπολογισμού και στο πλαίσιο των υφιστάμενων διαδικασιών θα μπορούσαμε ενδεχομένως για τα επόμενα 7 χρόνια να συστήσουμε ένα μηχανισμό που θα βοηθάει τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης. Αυτό είναι καθαρά και μόνο θέμα πολιτικής βούλησης. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχουν κριτήρια όπως παραδείγματο χάρη είναι διαφάνεια. Όμως δεν είναι δυνατόν σήμερα ένας υπάλληλος να αποφασίζει το τι θα γίνει ε, με την ελεύθερη δημοσιογραφική εργασία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να επιδείξουμε πολιτική βούληση και να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να στηρίξει τα μέσα ενημέρωση σε μια χώρα που γεωγραφικά βρίσκεται στην Ευρώπη. Ε, καταπιέζεται ε, από τη δημοκρατία, ζει έναν ελευθερία Άρα δηλαδή εδώ καλούμεθα να επιδείξουμε ε, αποφασιστικότητα για να βοηθήσουμε τα ελεύθερα μέσα ενημέρωση. Πρόεδρος, συνοψίζω τώρα και θέλω να επισημάνω ότι αυτό το πρόβλημα ε, τα πακέτα των ε, αιτήσεων που πρέπει κανείς να υποβάλει για να έχει πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό το πρόβλημα υφίσταται παντού. Όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι εντάξει μπορεί κανείς ε, να το δεχτεί σε μια δημοκρατία που δεν λειτουργεί σωστά η διοίκηση. Υποφέρουμε όλοι στα πολιτιστικά προγράμματα, υποφέρουμε όλοι από αυτό το γεγονός. Βέβαια αυτό οφείλεται ε, σε υπερβολικούς ε, κανονισμούς όπου υποτίθεται μερικοί είναι θεματοφύλακες για να μην χαθεί ούτε ένα, μία δραχμή, ένα σέντ στα, στις χορηγήσεις. Ο κύριος Μαρτίν είναι στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Ξέρει βέβαια ότι υπάρχουν ε, καταχρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτές τις υπερβολικά υπερβολικές ρυθμίσεις ε, που είναι σαν ε, το κρεβάτι του προκρούστη. Μας βάζουν εκεί και πρέπει να προσέχουμε και το τελευταίο σέντ στον πολιτιστικό μας τομέα μιλάμε για μικρά ποσά ή στις αδελφοποίησεις πόλεων. Εκεί δεν πρέπει να υφίσταται αυτή η τεράστια γραφειοκρατία. Όταν έχουμε μία γειτονική χώρα που άδεια αμφισβήτητα έχει δικτατορία, μπορεί κανείς να προσπαθήσει να βοηθήσει τους ανθρώπους, τους πολίτες της χώρας αυτής. Με λιγότερη γραφειοκρατία να βοηθάει τα μέσα ενημέρωσης. Με τα 200.000 ευρώ που σας δίνουμε βεβαίως δεν μπορείτε να ζήσετε, χρειάζεστε πολλά περισσότερα χρήματα. Πιστεύω πάντως ότι πρέπει να ε, προτείνουμε, γιατί σε τελική ανάλυση δεν έχουμε και τόσες πολλές δικτατορίες ε, στη γειτονιά μας, προτείνω λοιπόν να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, σε αυτή αυτή την ε, περίπτωση ε, για την ε, οποία γίνεται συνεχώς λόγος για πολιτικούς κρατούμενους, για την κυρία βεβαίως που κρατείται. Καλά, εντάξει, να αυτή την κυρία, αλλά υπάρχουν και εκατοντάδες άλλων κρατουμένων που υποφέρουν. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι μπορούμε να σας υποσχεθούμε κάτι συγκεκριμένο. Πάντως, αυτό που προτίθεμαι να κάνω και νομίζω αυτό εννοούσε και ο συνάδελφος κύριος Μάρτιν, εξ ονόματος της Επιτροπής, βέβαια θα κάνουμε κάποιες έρευνες και θα γράψω μια επιστολή προς την κυρία Άστον και θα την παρακαλέσω να σκεφτεί το κατά πόσον για αυτή την ειδική περίπτωση, εφόσον έχουμε δικτατορία στα πόδια μας, να συστήσουμε ένα ταμείο από το οποίο θα μπορεί κανείς ε, να ανακαλέσει κονδύλια. Βεβαίως, ε, στο τέλος θα χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία ε, και επίσης μπορεί και κανείς να αποδείξει θέματα ακροαματικότητας και θεαματικότητας. Κύριε Μιγκάλσκι, αν εσείς έχετε περισσότερες πληροφορίες, θα σας ήμουν ευγνώμων να μου δίνατε έγγραφα, τα στοιχεία σε γραπτή μορφή, να τα υποβάλω στην κυρία Άστον και να την παρακαλέσω να επιδείξει κάποια εφευρετικότητα. Δηλαδή, δεν έχουμε εδώ να κάνουμε με μια φυσιολογική κατάσταση. Έχουμε τη δικτατορία στα πόδια μας όπως σας είπα. Ε, και υπάρχει μια γειτονική χώρα που στηρίζει ε, αυτήν που μας ενδιαφέρει, όμως έχουμε και τον Πούτιν που στηρίζει τη Συρία. Εν πάση περιπτώσει, ε, θα με ενδιέφερε να έχω κάποια στοιχεία για να μην επιδείξω εραστεχνισμό. Ε, σας παρακαλώ λοιπόν να μου δώσετε τα στοιχεία, θα, συστήσω, θα συντάξω αυτή την επιστολή, θα παρακαλέσω βέβαια τους συναδέλφους να την υπογράψουν και αυτή η επιστολή, θα πάει στην κυρία Άστον να προσπαθήσει να διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχουν δυνατότητες να βοηθάει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, ε, σας ευχαριστώ κύριε Μιγκάλσκι που ήρθατε κι εσείς Πράγματι μερικές φορές ε, πρέπει κανείς να μας ε, ανοίξει τα μάτια. Σας ευχαριστούμε πολύ ε, και σας ευχόμαστε καλή ακροαματικότητα. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Χθε είχαμε τη συνεδρίαση των συντονιστών. Στείλαμε mail Δεν έχει υπάρχει τίποτα στα διάφορα. Επόμενη συνεδρίαση είναι 10 Ιουλίου στις 9 το πρωί. 10 Ιουλίου πρωί και μεσημέρι και στις, δηλαδή πρωί και απόγευμα και στις 11 Ιουλίου μόνο πρωί. Θα δούμε τώρα ανάλογα πώς θα διαμορφωθεί η ημερήσια διάταξη. Αν δεν χρειαστεί θα διαγράψουμε την ε, ε, τελευταία συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους διερμηνείς και τους Ρώσους ε, διερμηνείς. Ευχαριστεί η Πρόεδρος. Καλή όρεξη.